Επίση, Επίσης, καταφέραμε να εμποδίσουμε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για περιορισμό ε, του δικαιώματος επιστροφής χρονικά. Αυτό το καταφέραμε. Και μια σειρά από μέτρα ε, που πρέπει να γραφούν στο μαύρο κατάλογο. Δεν μπορώ να τα απαριθμίσω όλα γιατί δεν έχω χρόνο. Δεν καταφέραμε όμως σε αυτό το μαύρο κατάλογο να βάλουμε τα προϊόντα διτής ποιότητας που κυκλοφορούν με διαφορετική ποιότητα αλλά με την ίδια επωνυμία στα διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί κάποια μέλη αντιτάχθηκαν. Όλα αυτά όμως που καταφέραμε θα πρέπει να τα πετάξουμε στο κάλαθο των αχρήστων επειδή δεν πετύχαμε το τελευταίο. Παρόλα αυτά η ομάδα μου συνιστά υπερψήφιση και να φροντίσουμε στη ρήτρα αναθεώρηση που επίσης επιβάλαμε ε, στην επόμενη θητεία να το κοιτάξει και να αξιοποιηθεί για να λυθεί και αυτό το θέμα. Τα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές πραγματικά να επιβάλλονται παντού και απέναντι σε αυτή τη διπλή διαφορετική ποιότητα, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν καταναλωτές πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ή ποιότητας. Γι' αυτό ως σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλιστές και δημοκράτες θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για να καταργηθεί αυτό, γιατί είναι απαράδεκτο. Παρ' όλα αυτά αύριο θα υπερψηφίσουμε, γιατί πραγματικά πετύχαμε πολλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τη δική μου γενιά και για τους ανθρώπους από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όταν έπεσε το σύνδρομο παραπέτασμα. Θεωρήσαμε ότι ενώθηκε η Ευρώπη, αλλά για τα παιδιά μας θα είναι η θέση σε ισχύ της νομοθεσίας που απαγορεύει τις διαφορές ποιότητας. Το είδαμε να συμβαίνει. Ο κόσμος στην Ανατολική Ευρώπη ε, έχει ε, προϊόντα χειρότερης ποιότητας από ότι ο κόσμος στη Δυτική. Γι' αυτό το λόγο αυτός ο αγώνας κατά της ε, κακής ποιότητας των τροφίμων είναι πολύ εύστοχος. Έχει υποσχεθεί η Κομισιόν κάτι τέτοιο από το 2017. Το 2017 είπε ο κύριος Γιούνκερ ότι οι Σλοβάκοι δεν μπορούν να τρώνε προϊόντα χειρότερης ποιότητας. Δεν τους αξίζει κάτι τέτοιο να έχουν λιγότερο κακάο στη σοκολάτα τους και οι Ούγγροι δεν πρέπει να έχουν λιγότερο κρέας στο φαγητό τους. Ευχαριστούμε λοιπόν τους πολίτες που επεσήμαναν τα ζητήματα σε μας και ευχαριστούμε σε όσους έδειξαν διεθνή συνεργασία ε, κατά όσων μας παραπλανούν εδώ και χρόνια. Αυτή η νομοθεσία δεν είναι παρά ένα πρώτο βήμα ε, για να βελτιώσουμε την ισότητα και σε άλλους τομείς όπως τις γεωργικές ενισχύσεις. Για την ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Σελίμοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγα χρόνια αγόρασα online, μάλλον έκλεισα δωμάτιο σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο με καταπληκτική θέα, με πολύ ωραία έπιπλα και ήταν και τζάμπα σχεδόν. Πραγματικά δεν το πίστευα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Και πραγματικά όταν έφτασα εκεί, καλά έκανα και δεν πίστευα στα μάτια μου, γιατί πρώτον ούτε ξενοδοχείο ήταν, ένα γκαράζ ήταν, που κάποιο είχε κάνει ένα δωμάτιο, υποτίθεται που θα έμενα εγώ εκεί. Η νομοθεσία λοιπόν αυτή ακριβώς αυτό το στόχο έχει, να αποφεύγει τέτοια σενάρια στο μέλλον. Διότι αυτή είναι μια εμπειρία που έχουν ζήσει πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές και στην καθημερινή τους ζωή ε, η πρόταση αυτή το ε, απαγορεύει και είναι μια νίκη για τους καταναλωτές. Έχουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, πολύ σημαντικό, και ε, είναι και πάρα πολύ λογική η πρόταση για αυτό το επίμαχο θέμα της διαφορετικής ποιότητας των προϊόντων. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούμε, αλλά είναι καλό αυτό που πετύχαμε. Και επίσης δυσκολεύει σε αυτούς τους απατεώνες, ε, τους ε, μη σοβαρούς, να ε, σας εξαπατούν. Με τη διαφάνεια αυτή θα δείχνουμε ότι τα κριτήρια ταξινόμησης είναι ξεκάθαρα στο site και θα σταματήσουμε το να υπάρχουν ψευδείς αξιολογήσεις πελατών και αυτή η καταπληκτική θέα θα εξασφαλίζουμε να είναι πραγματικά καταπληκτική και θέα. Παρακαλώ να μην πέσουμε στην παγίδα ε, του να το επαναπέμψουμε το θέμα στην αρμόδια επιτροπή λόγω αυτού του επίμαχου θέματος της ποιότητα. Για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς το λόγο έχει ο κύριος Σύρντεβαν για ένα λεπτό. Ε, Κύριε ευχαριστώ ε, συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, καλό είναι που η Ευρωπαϊκή Ένωση αφοσιώνεται και ασχολείται με την προστασία των καταναλωτών και θέτει ευρωπαϊκού κανόνε και πρότυπα. Και καλό είναι που και το Κοινοβούλιο ω άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο είναι πιο αξιόπιστο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οποία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, άλλα ε, πρέσβευε και ήθελε για το δικαίωμα επαναχώρηση. Από ό,τι φαίνεται σε αυτό το νέο deal για τους καταναλωτές υπάρχει ένα πρόβλημα που ξέρουμε όλοι. Αυτή η διαφορετική ποιότητα, ας πούμε στη Γερμανία, πα με το παιδί σου στην Πολωνία και θες να του αγοράσει τα αγαπημένα του μπισκότα. Αυτά τα μπισκότα θα πρέπει ε, να έχουν βούτυρο και όχι φινικέλαιο, όπως έχουν τα ίδια μπισκότα στη Γερμανία. Αλλά δεν είναι η ίδια γεύση, ούτε η ίδια ποιότητα. Και αυτές είναι αθέμητες πρακτικές για μεγιστοποίηση του κέρδους και πλήττονται οι ε, καταναλωτές στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική και είναι καταναλωτές δεύτερης κατηγορίας. Ε, θα πρέπει να τερματιστούν αυτές οι πρακτικές στην κοινή και αλληλέγγυη Ευρώπη. Ευχαριστώ. <coughs> Για την ομάδα των Πρασίνων το λόγο έχει η κυρία Ρέντα για ένα λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πολλά, παρά τις καλές διατάξεις για τη διαφάνεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών, λείπει ένα βασικό κομμάτι από αυτή την νομοθεσία. Πλήρης απαγόρευση της διπλής ποιότητας των προϊόντων. Λυπάμαι που το κοινοβούλιο αυτό έχει χωριστεί όχι διολογικά, ε, αλλά γεωγραφικά και τα μέλη των δυτικών κρατών έχουν την εντύπωση ότι είναι αρκετά καλή η συμφωνία παρότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του της, ε, για την απαγόρευση της διπλή ποιότητα στο Κοινοβούλιο, ενώ τα κράτη τη Ανατολική Ευρώπη ζητούν καλύτερη συμφωνία. Η ομάδα των Πρασίνων δεν έχει ε, διαιρεθεί από αυτού. Πιστεύουμε ότι πρέπει οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζονται με ισότητα και αυτό αναμένουν και οι πολίτε. Δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσει λόγω του τόπου κατοικία και γι' αυτό να ε, αγοράζουν χαμηλή ποιότητα προϊόντα. Γι' αυτό ήρθε η στιγμή να το κάνουμε σωστό και να μην εγκρίνουμε τη συμφωνία του τριμερού διαλόγου που πέρασε βιαστικά και όπου το Κοινοβούλιο παρετήθηκε από την υπόσχεσή του στους πολίτες να απαγορεύσει τα προϊόντα διπλής ποιότητας. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει ο κύριος Γκουόγκα για 1,5 λεπτό. Thank you, President, Commissioner, Rapporteur. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Συγητή. Είναι σημαντική ημέρα. Ε, παρόλα Παρόλε τι προσπάθειε, είναι δύσκολο να επιτευχθεί όπω φαίνεται μια συμφωνία που δεν θα έχουμε διακριτική μεταχείριση. Κάθε εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, είδαμε διάκριση των περιφερειακών χωρών στο πακέτο για την κινητικότητα και τώρα θέλουμε να μεταχειριζόμαστε ανθρώπου διαφορετικά, δίνοντά του προϊόντα χρησιμοποιημένα. Αυτό του δίνουμε, δεύτερη κατηγορία. Γιατί του μεταχειριζόμαστε διακριτικά. Και α το παραδεχτούμε. Θέλουμε τι, να αποτύχουν όλοι δεν θέλουμε ίδια ποιότητα προϊόντων για όλους, ναι. Ας μην τα παρατάμε, ας συνεχίσουμε τη μάχη και ας κερδίσουμε αυτή τη μάχη ώστε όλοι να έχουμε μια δίκαιη Ευρώπη. Αυτό ζητάμε, ίσα δικαιώματα, ίση Ευρώπη. Όλοι να κερδίζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σενάλοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ε, ο συμβιβασμό αυτός λέγει ότι ε, βελτιώνει την κατάσταση των καταναλωτών και αν δεν εγκριθεί ε, θα πρέπει να περιμένουν άλλο ένα χρόνο οι καταναλωτές. Ναι, και αυτό τώρα τι είναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά τα δικαιώματα των μεν ενισχύονται και των δε ε, επιδεινώνονται. Δεν υπερψήφισα και έκανα και τροπολογία που ε, ζητάει συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται να φύγουμε από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων εάν δεν ε, καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα και να έρθουν να πούνε στους ε, πολίτες των χωρών μας ότι σταματάει αυτή η αθέμητη πρακτική. Γιατί είναι αθέμητη πρακτική όταν έχει την ίδια μάρκα το ίδιο προϊόν αλλά διαφορετική ποιότητα ανάλογα με το που πωλείται. Αγαπητοί συνάδελφοι, μην αλλάξετε τη γνώμη ε, που εκφράσαμε ήδη στο Κοινοβούλιο. Όλοι συμφωνήσαμε και όλοι είπαμε ότι θέλουμε να απαγορευτεί η διπλή ποιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το αξίζει. Το λόγο έχει η κυρία Χαράντσοβα για λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή είναι η τελευταία μας ολομέλεια. Μας δόθηκε η ευκαιρία και πράγματι έπρεπε να θέσουμε τέλος της συζητήσεις για την περιεκτικότητα κακάο σε σοκολάτες. Εγώ ως ε, βουλευτής της Τσεχική Δημοκρατίας είμαι απογοητευμένη από το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να ψάξω να βρω από δύο πομπέο τράγο σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι η πίεση από τα κράτη-μέλη ή η πίεση από τις επιχειρήσεις που γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ με προϊόντα κακή ποιότητας. Αλλά ξέρουμε ποιο πληρώνει τελικά την ύφη. Είναι οι καταναλωτέ ε, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ σκληρή αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων, των κατοίκων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και τα πράγματα είναι ανωκάτω και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Ε, τουλάχιστον έχουμε μια πρόταση που προσπαθεί κάτι να κάνει, αλλά δεν είναι παρασυμβολική αυτή η νομοθεσία. Δεν θα φέρει επαρκές αποτέλεσμα. Δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί και να προστατεύσει πραγματικά τους ανθρώπους από τις εθέμητες πρακτικές. Το αφήνουμε δηλαδή στους παραγωγούς. Ε, τους, το κάνουμε ε, δώρο το να μπορούν να προσφέρουν προϊόντα διπλής ποιότητας ε, και να λένε ότι είναι διαφορετικές οι γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τους συνεδρούς αύριο να υποστήριξουν τις δικές μας τροπολογίες και να θέσουμε τέλος σε αυτή την πρακτική δύο κατηγοριών καταναλωτών. Ευχαριστώ. Κυρία Χαραντσόβα, έχετε μια μπλε κάρτα από την κυρία Σόντροβα. Τη δέχεστε? Ναι. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι τη συναδέλφο. Δεν θεωρείτε, κυρία Χαράντσοβα, ότι υπερβάλλεται κάπως ε, στο πώς διατυπώνετε τα πράγματα. Εδώ και χρόνια ξέρετε ότι υπήρχε διπλή ποιότητα στα τρόφιμα, αλλά και σε άλλα αγαθά. Και για χρόνια ε, έπρεπε να σταματήσει αυτή η αθέμητη πρακτική και μόλις αυτή η Κομισιόν, αυτό η Επίτροπος κατάφερε επιτέλους να κάνει κάτι, όχι ο κύριος Γιούνκερ, οι Ευρωβουλευτές το κατάφεραν, ε, οι ακτιβιστές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε. Αγαπητοί Αγαπητή συνάδελφε, όπως σας είπα είμαι απογοητευμένη από το αποτέλεσμα. Ναι πράγματι το κοινοβούλιο αυτό αγωνίστηκε εδώ και μερικά χρόνια για να θέσει τέλος σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Αλλά το κείμενο αυτό δεν είναι το κείμενο που ήθελε το Κοινοβούλιο, ούτε η θέση της Επιτροπής μου. Δεν αγωνίστηκα γι' αυτό, γι' αυτό είμαι απογοητευμένη. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κονέτσνα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από τότε που μας υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα καταργηθεί διπλή ποιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σημερινό κείμενο τι κάνει, το αντίστροφο. Διατηρεί το status quo, αυτό το όνειρο. Και μάλιστα προωθεί ε, τη θέση της μη εκλεγμένης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά τον τελευταίο τριμερή διάλογο έγιναν διάφορες παρασκηνιακές συνεννοήσεις, περίεργες. Τι είναι αυτή η διατύπωση. Ε, θα το πάρουν πολύ άσχημα οι πολίτες στην τσεχική δημοκρατία αν περάσει έτσι αυτό το κείμενο. Από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιβάλλει κάποιες επίμαχες ε, διατάξεις και υποχρεώσεις και από την άλλη οι δυτικές χώρες ε, μας κάνουν dumping και μάλιστα δεν το κρύβουν κιόλας. Ε, δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα μετά η παρηγοριά παρά να εγκρίνει ο καθένα την εθνική του νομοθεσία. Γι' αυτό υποστηρίξτε παρακαλώ τις τροπολογίες μας για να επανέλθουμε ε, στον συμβιβασμό και να σταματήσει αυτή η επονίδιστη ε, πρακτική. Το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες δεν έχει νόημα γιατί οι πολίτες δεν είναι όλοι ίδιοι. Έχει κυρία Σούιτσα για λεπτό drago mi Όσον αφορά αυτή την οδηγία, περιλαμβάνει τη προϊόντα διπλής ποιότητας και τέθηκαν πολλά ερωτήματα στην Κομισιόν όσον αφορά τη διακριτική μεταχείριση και τη διπλή ποιότητα. Η απάντηση της Κομισιόν προς εμένα ήταν ότι τα αποτελέσματα έδειχναν ότι οι καταναλωτές έχουν διαφορετική γεύση. Εγώ έχω την υποστήριξη 44 ευρωβουλευτών. Επι... Πραγματοποίησα και μια μελέτη και πρότεινα και ενωσιακή νομοθεσία να υπάρξει ώστε να δοθεί τέλος σε αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Έγινε συζήτηση στην Ολομέλεια μαζί με τον ε, συνάδελφο Σόιντροβα από την Τσεχική Δημοκρατία για τα αποτελέσματα μετά από τη δοκιμή γερμανικών, κροατικών και τσεχικών προϊόντων. Ο κύριος Γιούνκερ πρότεινε μια νέα συμφωνία. Και δεσμεύτηκε από αυτό. Η θέση του Κοινοβουλίου ήταν σαφής. Δείξαμε ε, στην ψηφοφορία μας το Σεπτέμβριο ότι το κείμενο όπως χρησιμοποιήθηκε στον τρίλογο δεν ήταν ικανοποιητικό. Εγώ υπέβαλα τροπολογίες με στόχο να διασφαλίσει τη ίδια ποιότητα για όλους τους πολίτες και απευθύνω έκκληση προς τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτές τις τροπολογίες γιατί προσπαθούμε να πολεμήσουμε αυτή την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Ζητώ συγγνώμη, ε, θα, συγγνώμη, θα λυπηθώ εάν θα επικραθώ αν δεν γίνουν δεκτές οι τροπολογίες αυτές θα εμβαθύνουν τις διαφορές μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ογιούνκερ ο ίδιος είχε πει εδώ ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπνέει και με τους δύο τις πνεύμονες εξίσου. Παρακαλώ, μην το ξεχνάτε ψηφίζοντας αύριο. Λεπτό το λόγο έχει κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαφές ότι οι οδηγίες αυτές έπρεπε να τροποποιηθούν. Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να τροποποιήσει τέσσερις οδηγίες, δικαιώματα καταναλωτών, αθέμητες εμπορικές πρακτικές, διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις, ε, τιμολόγηση κτλ. Βεβαίως, οι περισσότερες αλλαγέ γίνονται στις δύο πρώτες οδηγίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά να έχουμε την ίδια ποιότητα στα προϊόντα μας παντού στην εσωτερική αγορά. Να σεβόμαστε όλου του καταναλωτέ, εξίσου εξαρτήτως χώρα στην οποία ζουν. Είναι καλέ. Ε, οι αλλαγές που έχουν γίνει και δεν μπορούμε να τις παραγνωρίσουμε. Σκέφτομαι εδώ το δικαίωμα των καταναλωτών να αποσυρθούν από τη σύμβαση να, να αλλάξουν γνώμη, να αποζημιώνονται. Βεβαίω ο συμβιβασμό δεν φτάνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε εμεί. Παράδειγμα, ε, είναι πιο σαφής για τη διαφορετική ποιότητα του ίδιου προϊόντος. Ε, μπορεί να έχει αλλάξει το άρθρο 6 της οδηγίας, αλλά ε, ε, εισάγονται κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες έχουν αποδυναμώσει πάρα πολύ την ισχύ του άρθρου 6. Βεβαίως υπάρχει ρήτρα αναθεώρησης ε, και αυτή θα μπορούσε να είναι η λύση. Τώρα είμαστε και λίγοι εδώ. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να καθίσουν και να το σταθμίσουν. Ζυγίστε το. Είναι καλύτερο να καταψηφίσετε ή να υπερψηφίσετε. Όλοι το ίδιο θέλουμε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ακράδαντα ότι η οδηγία αυτή στο σύνολό τη ε, είναι ευεργετική και επωφελής για τους καταναλωτές. Πραγματικά θα τους προστατεύει από αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Και αυτό είναι θέμα που υπάρχει παντού στην Ευρώπη, όπως και επιθετικές πωλήσει ε, ή ε, ψευδείς αξιολογήσεις πελατών, υποτίθεται, παραπλανητική διαφήμιση ή ψευδείς ε, και πλαστές ε, εκπτώσεις. Και υπάρχουν δύο πράγματα που είναι ιδιαίτερα θέμητα μεταξύ αυτών. η επιτυχία ε, αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, υπιστώνεται σε Τσέχους. Και ευχαριστώ την Επίτροπο Γιούροβα και την Μάνδρια Μαρέτσκα, πρώην Υπουργό, που έχει ανακοινήσει αυτό το θέμα στο Συμβούλιο και έχει επιμείνει πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την κατάρτιση της ε, πρότασης αυτής. Ε, το ξέρω ότι δεν είναι τέλεια. Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους που το είπαν. Και επίσης συμφωνώ ότι θα μπορούσαμε και θα πρέπει να προχωρήσουμε και να έχουμε ένα σαφή ορισμό. Όλα αυτά είναι ωραία. Αλλά μετά από μία διετία ε, είναι πολύ αργά να ξαναγυρίσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν κάποια σημεία που αν δεν ε, λειτουργούν θα τα δούμε τη στιγμή της αναθεώρησης, γιατί η οδηγία προβλέπει αναθεώρηση. Υποστηρίζω τις τροπολογίες αυτές, αλλά πιστεύω ότι καλό θα ήταν να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπόρζεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ εδώ και έξι χρόνια όταν άρχισα να ασχολούμαι με το πρόβλημα της διπλής ποιότητας μου φαινόταν απίστευτο ότι σήμερα θα υπήρχε ένα νομοθέτημα που απαγορεύει αυτή την άδικη πρακτική. Αυτό είναι αποτέλεσμα έρευνας, συστάσεων, συζητήσεων ε, έξι ετών. Κανείς τώρα πια δεν μπορεί να πει ότι οι Κροάτες ή οι Βούλγαροι έχουν, ε, τρώνε τροφές που δεν είναι τόσο υγιείς, υγιεινές ή ότι είναι χαμηλότερη ποιότητα η τροφή τους. Για μένα και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή είναι μια πολύ συγκινητική κατάσταση. Μας κάνει να νιώθουμε πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Πολύ σωστά το Κοινοβούλιο δείχνει ότι δεν υπάρχει διάκριση Ανατολής Δύσης, ότι είμαστε μία Ευρώπη, ότι μπορούμε και οφείλουμε όλοι να είμαστε ίσοι. ότι δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοιου είδους πρακτικές. Η, ισότητα είναι, είναι το μήνυμα που στέλνουμε στην Ευρώπη. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι απογοητευμένο με το σύμβασμο που επιτύχαμε στον Τριλόγο. Ο σύμβασμος αυτό θεωρώ δεν θα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη διπλή ποιότητα των τροφίμων στην πρακτική. Θα καταλήξουμε σε διαφορετικέ ερμηνείε. Για παράδειγμα, θα γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τις μάρκες, τι περιέχουν και όσοι θα συνεχίσουν να παράγουν προϊόντα διπλής ποιότητας ε, θα γελούν μαζί μας. Ε, θέλουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ελπίζω το Συμβούλιο να μην τιμωρήσει κανέναν τελικά αν περάσει η τροπολογία μας και να βελτιώσουμε τον ορισμό των αθέμητων πρακτικών. Είμαι υπέρ του να λέμε σαφώς ότι τα τρόφιμα διπλής ποιότητας αποτελούν αθέμητη πρακτική και τέλος. Αντί να έχουμε μια λίστα εξαιρέσεων προστατεύοντας τους μεγάλους ομίλους ε, που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική ε, και που βρίσκουν ε, αγορά προϊόντων χαμηλή ποιότητα στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση, αλλά δυστυχώ η Τσεχία υποστήριξε τη συμβαστική. Είναι προσβολή προ του πολίτε τη του ίδιου. Και εγώ θα ήμουν ευγνώμων αν εγκρίνατε τι ε, τροπολογίε που υποβάλαμε αύριο για να έχουμε την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι αν παράγει κανείς διπλή ποιότητα ε, θα θεωρείται ότι εφαρμόζει αθέμητες πρακτικές. Δεν πρέπει να κοιτάμε το πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές καθόλου. Οπότε Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί 7 αιτήματα. Θα κάνω και τα 7 αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Μπούσο Κρίστιαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ε, αποτελεσματικής εταιρικής ε, εμπορικής δραστηριότητας και προστασίας των καταναλωτών. Για πρώτη φορά έχουμε συγκεκριμένες αναφορές σε διπλά πρότυπα και τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν μέτρα. Αλλά θα πρέπει να, έπρεπε να είμαστε πιο φιλόδοξοι και με καλύτερες προδιαγραφές. Οι πρακτικές αυτές υπονομεύουν την ίδια την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στον κέντρο ε, ευρωπαϊκών και ανατολικοευρωπαϊκών κρατών, εμπιστοσύνη στην εσωτερική μας αγορά. Θέλω να υποστηρίξουμε την τροπολογία της συναδέλφου Ρόζα Τούν που ψηφίστηκε αρχικά ε, στην Επιτροπή ΥΜΚΟ και έτσι θα βελτιωθεί ακόμα η κατάσταση. Το λόγο έχει η κυρία Ζωάνα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, ε, υπάρχουν τα διπλά στάνταρ ε, και ε, οι προδιαγραφές αυτές. Ακούσαμε τα διάφορα επιχειρήματα και ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τη διπλή ποιότητα, για τις διπλές προδιαγραφές, ό,τι και αν πιστεύει κανείς για τα γούστα των Ανατολικοευρωπαίων που υποτίθεται ότι είναι διαφορετικά από εκείνα των Δυτικών πρέπει να σας πω κυρία Επίτροπε ότι έχουν βαρεθεί έχουν μπουχτίσει οι Ανατολικοευρωπαίοι να τους ταΐζουν ε, τέτοια κακά προϊόντα και τρόφιμα ε, κατώτερης ποιότητας ε, και χειρότερης ποιότητας το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα να αγοράζουμε αυτοκίνητα κατώτερης ε, ποιότητας που είναι πασιφανές ότι είναι χειρότερα από όσα κυκλοφορούν στη Δυτική Ευρώπη. Ολόκληρο το ανατολικό μπλοκ 30 χρόνια και παραπάνω ε, ε, έχει συνηθίσει να υπάρχει ποιότητα για όλους, την ίδια ποιότητα. Δεν μπορούμε πια να γελιόμαστε. Ε, δεν επιτρέπεται να θεωρούν κάποιοι άλλοι ότι έχουμε διαφορετικά πρότυπα από τους δυτικοευρωπαίους. Πρέπει, πρέπει και εμεί να έχουμε τα ίδια προϊόντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η προστασία των καταναλωτών απαιτεί να μην υπάρχουν διπλά στάνταρτς να μην υπάρχει η έννοια της διπλής ποιότητας και έτσι να έχουμε τη διάκριση εις βάρος των καταναλωτών ιδίως στην ανατολική ευρώπη. ταυτόχρονα προστασία των καταναλωτών σημαίνει προστασία του εμπορικού σήματος προστασία της εμπορικής επωνυμίας ιδίως των επιχειρήσεων που είναι εντός ευρωπαϊκής ένωσης έναντι αθέμητων πρακτικών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών και αυτό ισχύει ιδίως για τα ελληνικά προϊόντα τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και τα οποία χρησιμοποιούν τον διακριτικό τίτλο μακεδονικό όπως είναι μακεδονικό κρασί μακεδονικός χαλβάς και υφίστανται σήμερα ένα αθέμητο ανταγωνισμό από την πλευρά των σκοπίων που χρησιμοποιούν και αυτά την έκφραση μακεδονικός με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τεράστια πρόκληση και ταυτόχρονα σύγχυση. γι' αυτό κυρία επίτροπε κυρία Γιουρόβα, απαιτείται η ευρωπαϊκή επιτροπή να στηρίξει τα ελληνικά προϊόντα τα οποία είναι κατοχυρωμένα εδώ και χρόνια και τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και φέρουν τον τίτλο μακεδονικό. είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει η κομισιόν να το δει. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, για τη Σλοβακία και τις άλλες χώρες Ανατολικής Ευρώπης, το θέμα της διπλής ποιότητας, διαφορετικής ποιότητας των προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έχει αποδειχθεί ότι πολλές εταιρείες ε, διαθέτουν προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα, αλλά με διαφορετικά συστατικά και συνήθως χαμηλότερης ποιότητας. δύσκολο θα καταλήξουμε συμφωνία για την πρόταση αυτή, γιατί δεν είναι καλή. Και εκπλήσωμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέτει προθεσμία μία ακόμη διετία για την αξιολόγηση της κατάστασης. Και δεν ξέρω αν τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει απαγόρευση τέτοιου προϊόντο που είναι διαφορετικής ποιότητας. Γνωρίζουμε την ύπαρξη τέτοιων εμπορικών πρακτικών και οι πολίτε, ειδικά των δικών μα χωρών, είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Θα καταθέσω δύο τροπολογίε που προτείνουν την απαγόρευση τέτοιων πρακτικών. Γιατί αν έχουμε κοινή εσωτερική αγορά, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πολίτης μιας χώρας ε, μέλους που σχετικά πρόσφατα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ζωτική σημασία να μην έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά και διαφορετικές ποιότητες για τα ίδια προϊόντα ανάλογα με το που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλη νίκη για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες που ζητούμε αυτό το θέμα στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία και θα ήθελα να συγχαρώ τους δύο συναδέλφους για, την, ε, για το πόνημά τους και κυρίως ευχαριστώ την Όλγα γιατί χάρη στη δική της πρωτοβουλία συζητάτε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καμία λογική δεν υπαγορεύει σε μια ενιαία κοινή αγορά να μην έχουμε ενιαίες προδιαγραφές και πρότυπα για τα προϊόντα που διατίθενται με το ίδιο εμπορικό σήμα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε διαφορετικές ποιότητες για το ίδιο προϊόν. Α, τι ελεύθερη διακίνηση ε, εμπορευμάτων και υπηρεσιών έχουμε. Έχουμε πολύ επιλεκτική τέτοια διακίνηση. Γι' αυτό καλώ τις βουλγαρικές αρχές ε, να ενσωματώσω το συντομότερο δυνατό αυτή την οδηγία. Γιατί μετά από 10 χρόνια δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Κάνω Ευχαριστώ πολύ, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες διατάξεις που συζητάμε στην έκθεση απλούστατο ακυρώνουν όλη τη δουλειά που έκανα εγώ με την Όλγα Σετάνοβα ε, και με άλλους συναδέλφους τα τελευταία δύο χρόνια με την έκθεση που αφορούσε τα διπλά τα, αυτά πρότυπα. Ε, οι Ρουμάνοι και άλλοι κατανοτές Ανατολικής Ευρώπης διορτώνται τι κάνει η Ευρώπη για μένα. Γιατί η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαφορετικά τους ε, πολίτες βλέποντας ότι οι αξίες της Ένωσης θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους γιατί η Ευρώπη λοιπόν δεν μας αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο λένε οι Ανατολικοί. Δεν είναι δίκαιο έναντι των πολιτών που ψηφίζουν, μας ψηφίζουν και που μας στέλνουν εδώ. Διότι έχουν εμπιστοσύνη, διότι πιστεύουν ότι εμείς θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους. Όμως υπάρχουν τα συμφέροντα των μεγάλων εμπόρων, των μεγάλων εταιριών, αλλά είναι ντροπή που Επί Ρουμανική Προεδρία, οι Ρουμάνοι αντιμετωπίζονται σαν πολίτε δεύτερη κατηγορίας διότι από ό,τι φαίνεται δεν γνωρίζουν ε, τι είναι γραμμένο στα διάφορα έγγραφα. Λοιπόν, τελικά τους δίδονται, ε, μοιράζονται τα προϊόντα τα, ανάλογα με την γεωγραφική ε, περιοχή που μοιράζονται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποιος από μας θα προτιμούσε ένα προϊόν το οποίο να είναι παραφτιαγμένο ένα παγωτό που είναι φτιαγμένο από διαφορετικά ουσιαστικά, ε, συγγνώμη, από διαφορετικές ουσίες, με διαφορετική κρέμα από αυτή που αναφέρεται στο περιτύλιγμα. Αλλά βλέπουμε αυτό να συμβαίνει συνέχεια. Έχουν διαφορετικές ουσίες κάποια ποτά από χώρα σε χώρα, αναψυχτικά και αυτά θα πρέπει να τα εμποδίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο, την κυρία Σενάλοβα και τους άλλους συναδέλφους που μάχονται για ισότιμα δικαιώματα για όλους. Αυτή η διπλή ποιότητα δεν μπορεί να υφίσταται στην Ευρώπη. Είναι κάτι αντίθετο με τους κανόνε ενιαία αγορά. Διότι δεν, δεν πρέπει να έχουμε δύο κατηγορίε Ευρωπαίων. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να εμποδίσουμε αυτή τη διπλή ποιότητα. Εγώ υποστηρίζω τις τροπολογίες Δυστυχώ, η τσεχική δημοκρατία υποστήριξε το συμβιβασμό που καθιστά πιο αόριστο τον ορισμό και δεν βελτιώνει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στην τροπολογία σα ζητώ να τις υποστήριξετε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Εξ της Επιτροπής το λόγο έχει και πάλι η Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτά, ξαφνικά σκέφτηκα δεν μιλάω τσεχικά, τη μητρική μου γλώσσα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Για έναν πολύ εύλογο λόγο, για να δείξω τη στάση που έλαβα στο θέμα της διπλής ποιότητας προϊόντων. Γιατί είμαι κάτοικος της Τσεχίας και ως τέτοια νιώθω οργή όταν διαπιστώνω ότι κάποια εμπορεύματα στη χώρα μου κυκλοφορούν σε χαμηλότερη ποιότητα από ό,τι τα ίδια προϊόντα σε άλλες χώρες. Έκανα περιοδία σε πολλά γεωργικά επιμελητήρια χωρών μελών και άκουσα πολλές ε, αμφιβολίες ε, για το κατά πόσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, για το κατά πόσο είναι υπαρκτό αυτό το πρόβλημα. Άκουσα όμως ταυτόχρονα και τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Σέχναλοβα, η κυρία Μπόρζαν και άλλοι, εδώ και χρόνια εμ, επισημαίνουν το πρόβλημα που δεν είναι από κύμα της φαντασίας α, κάποιου χασομέρι που δεν έχει τι να κάνει και επινοεί προβλήματα. Όχι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το γεγονός ότι σήμερα καταθέτουμε οδηγία που αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτού του προβλήματος, την οδηγία για τις ε, αθέμητες εμπορικές πρακτικές, νομίζω ότι συνιστά ένα βήμα προόδου. Ε, εξέτασα ε, προτάσεις 8 χωρών για τις ε, διάφορες πρακτικές που ισχύουν σε χώρες. Έγιναν διαβουλεύσεις με την βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και μου είπαν ότι θα πρέπει να μπερδεύουμε διαφορετικά πράγματα, ότι δεν είναι το πρόβλημα σοβαρό, ότι δεν θα πρέπει να εγκύψουμε σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό ε, πέρασε σε μια δεύτερη έρευνα επιλεγμένων προϊόντων από τα κράτη-μέλη και διαπίστωσα ότι 20 με 30% των προϊόντων αυτών παρουσιάζουν αισθητέ διαφορές στην ποιότητα ανάλογα με τη χώρα στην οποία διατίθενται. Γι' αυτό και είπαμε θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων ή των επιθεωρήσεων. Δεν πρόκειται να επιβάλλουμε στα τα κράτη-μέλη ε, τι επιθεωρήσει θα πρέπει να κάνουν και με τι δειγματοληψία θα πρέπει να κάνουν τη σύγκριση των προϊόντων που διατίθεται στην αγορά. Αλλά τώρα έχουμε καταλήξει σε μια συντονισμένη μέθοδο και πιστεύω ότι με τη μεθοδολογία που προτείνουμε σήμερα μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματά σας ότι κυκλοφορούν σοκολάτες ή παγωτά διαφορετικής ποιότητας. Ε, ακριβώς σε αυτά τα πράγματα που μας ενοχλούν επικεντρωθήκαμε, γιατί σίγουρα ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους ελέγχους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται σωστή δειγματοληψία και να ασκούνται να εφαρμόζονται τα κείμενα. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε χαμηλότερο ποστό κακάο από ό,τι προβλέπετε για τη σοκολάτα, το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται παραποιημένο, νοθευμένο και να αποσύρεται από την αγορά τέτοια προβλήματα θα διορθώσει η οδηγία, προβλήματα που ενοχλούν τον ε, καταναλωτή και θα ενισχύσουν έτσι την εμπιστοσύνη του στις επιθεωρήσεις και στους ελέγχους της αγοράς. Πιστεύουμε ότι θα, θα δείξουμε κουράγιο και θα εφαρμόσουμε την οδηγία πιστά. Κύριε Ποσπίσιλ, μας κατηγορήσετε ότι οι νομικές έννοιες είναι υπερβολικά γενικές και αόριστες. Μα πολλές νομοθετικές πράξεις ε, έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Από τη στιγμή που έχουμε διαφορετικές ποιότητες, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το ζήτημα της ποιότητας. Γιατί δεν μιλούμε μόνο για τρόφιμα, μιλούμε γενικώ για προϊόντα. Και το γεγονός ότι εγώ ως επίτροπος αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, είμαι υποχρεωμένη να καλύψω ε, ένα ευρύ φάσμα προϊόντα και τα καλλιτικά, τα αρώματα, τα αυτοκίνητα, δομικά υλικά και τρόφιμα. Είναι μεγάλο το φάσμα των προϊόντων. Γι' αυτό και θα πρέπει να ορίσουμε κάποιο τρόπο τι εστί αθέμητη εμπορική πρακτική. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις. και τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν επιλογή των δειγμάτων ε, θα ασκήσουν τον έλεγχο και θα επιβάλλουν και κυρώσεις ε, ενδεχομένως αναπερίπτωση. Ξέρω ότι στην πατρίδα μου ο αρμόδιος Υπουργός Γεωργίας θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και οι αρχές επιθεώρησης αγοράς ήδη έχουν ετοιμαστεί για να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή στην εθνική νομοθεσία και να ισχύσει το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει και κάτι άλλο. Πριν από 1,5 χρόνο δεν είχαμε τέτοια ευαισθητοποίηση και τέτοια ενημέρωση του καταναλωτή. Ε, φαίνεται ότι ο καταναλωτής ενεργοποιείται όλο και περισσότερο. Αλλά σήμερα, ακόμη και αυτοί που ε, έχουν απλώς κάποιες ε, υποψίες, αλλά όχι αποδείξεις, ακόμη και ενεργισμένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να ελέγξουν ότι ο ίδιος παραγωγός διαθέτει με το ίδιο εμπορικό σήμα το προϊόν, αλλά με διαφορετικές ποιότητες. Δεν μπορούν οι καταναλωτές να τα ελέγξουν αυτά. Θα πρέπει όμως οι ελεγκτές να εξασφαλίσουν αυτόν τον έλεγχο. Και σε περίπτωση που υπάρχει διπλή ποιότητα για το ίδιο προϊόν θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ο παραγωγός. Η διαφορετική ποιότητα δεν δικαιολογείται και ελπίζω ότι οι επιθεωρητές θα εντοπίσουν τέτοια προβλήματα και θα τα διορθώσουν. Και για αυτούς που θα, επι... θα προτιμούσαν πιο αυστηρή νομοθεσία, τι να σας πω, καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό, γιατί μερικές χώρες ήταν κατά της οποιασδήποτε ρύθμισης. Εγώ προσπάθησα με μια ενδιάμεση λύση να έχουμε μια σύγκληση απόψεων και να εξαλείψουμε τελικά διαφορετικές ποιότητες ε, προϊόντα με το ίδιο εμπορικό σήμα. Πιστεύω ότι έτσι θα, θα αποκαταστήσουμε μια ε, πραγματικά εύρυθμη εσωτερική αγορά. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και των λιανεμπόρων. Μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για τα προϊόντα. Επίσης προβλέπουμε και μια ρήτρα αναθεώρησης και να δούμε αν είναι κατάλληλη αυτή η νομοθεσία, αν είναι αποδοτική και αν θα πρέπει να δοθεί κάποια συνέχεια και αν διαπιστώσουμε κάποια κενά ή αδυναμίες στην τρέχουσα νομοθετική πρόταση, στο μέλλον η, αναθεώρηση, η αναθεωρημένη πρόταση θα είναι πιο αυστηρή. Πάντως, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε, γιατί αν αποσύρουμε τώρα την νομοθετική πρόταση, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο μελλον η αναθεωρημενη προταση θα έχουμε γυρίσει 1,5 χρόνο πίσω ουσιαστικά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε ε, στο πρόβλημα και να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, ε, χρησιμοποίησα όλη τη δημιουργικότητα, όλη την ευρηματικότητά μου, αλλά και την οργή που ένιωθα ως καταναλώτρια, για να ε, καταλήξω σε αυτή την πρόταση. Και πιστεύω ότι ορίμασαν οι περιστάσεις και ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να καταθέσω τη σχετική νομοθετική πρόταση και να προβλέψω και μία ενδεχόμενη αναθεώρησή της στο μέλλον. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση και η λύση δεν είναι να πούμε ότι είναι μία άλλη απόδειξη του χάσματος Ανατολής και Δύσης, ότι υπάρχουν διαφορές και ιδού η απόδειξη. Είμαι κατά αυτής της άποψης δεν θα πρέπει ε, να ε, αντιμετωπίσουμε την Ανατολική Ευρώπη ως ε, το σκουπίδο τενεκέ της Δυτικής Ευρώπης. Είμαι κατά αυτής της προσέγγισης και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση. Αυτά. Ευχαριστώ. Ελπίζω να εγκρίνεται αυτή τη συμβαστική λύση. Ευχαριστώ μεγάλο θέμα, αλλά 90% των παρεμβάσεων αφορούσαν μόνο ένα θέμα και συμφωνώ με αυτά που είπατε πολλοί από εσά για την διπλή αυτή ποιότητα και γι' αυτό πετύχαμε πολλά, θα έλεγα, πάνω σε αυτό. Είναι ρηξικέλευτη η συμφωνία αυτή για την διπλή ποιότητα, αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω γιατί οι συνάδελφοι σκοτώσουν όλη τη συμφωνία συμπεριλαμβανομένων των πάντων, διότι δεν πετύχαμε το ανέφικτο αίτημα να περάσει. Απλούστα το δεν είναι βιώσιμο να απαιτούμε το ίδιο σε όλες τις χώρε. Υπάρχουν διαφορετικά γούστα σε κάθε χώρα διαφορετικέ πρωτεσίλε σε κάθε χώρα και δεν είναι πάντα χειρότερα, τα συστατικά είναι διαφορετικά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Coca-Cola. Στο Ηνωμένο Βασίλειο φτιάχνεται με ζαχαροκάλαμο. Στο Βέλιο και στη Γαλλία με ζα... από ζαχαρότευτλα. Ε, ποια είναι η διάκριση εκεί. Ποιο χάνει τελικά το προϊόν που του αρέσει από τη βιομηχανία που θέτει στη χώρα του. Καταλαβαίνω τι ανησυχίε σα για την Ανατολική Ευρώπη. Αλλά στην περίπτωση ε, ε τη έχουμε τα όσο μπούκο. Είναι γλυκόζι που παράγει στην Ανατολική Ευρώπη. Το θέμα είναι ποιο είναι το καλύτερο προϊόν και ποιο είναι αντικειμενοδιάκη. Αν περάσει αυτή την τροπολογία, θα πρέπει αυτό να το κάνουμε για κάθε προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκατομμύρια εκατομμυρίων προϊόντων. Αυτό είναι ανέφικτο. Επίση, δεν είναι δυνατόν να περάσει αυτή την τροπολογία και να πάμε πίσω στι διαπραγματεύσει. Δεν θα υπάρξει διαπραγματευτική τράπεζα. Το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέσαν σαφέ ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και έκαναν πολλά. η ώρα Πέρασε η ώρα μάλλον και θα πρέπει να σαφέ για αυτού ότι δεν έχει νόημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει οτιδήποτε, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική θέση. Θα σημαίνει στο τέλο δεν θα έχουμε καμία συμφωνία. Και μετά θα χάσουμε τα εξή. Αυτά που πετύχαμε όσον αφορά τη διπλή ποιότητα, όσον αφορά τη διαφάνεια ε, διαβαθμολόγηση, το δικαίωμα απόσυρση, απαγόρευση, ε, απαγόρευση ψευδών πωλήσεων, σύγκριση υπηρεσίε για σύγκριση τιμών και διαφάνεια εκεί και τη δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσει. Α μην τα πετάξουμε όλα αυτά και πριν κλείσω, ευχαριστήσω εκείνους στο γραφείο μου που έγραψαν Κάμερον Σμιθ, ε, Τζέι Ντέιβις και Άλεκ Τζοφ. Ευχαριστώ πολύ που συνεργάστηκαν. Έληξε η ψηφοφορία, θα διεξαχθεί αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά στην έκθεση της κυρίας Αγιούζο με θέμα διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλωσίδα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει η κυρία Αγιούζο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερω που μετά από 20 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τελευταία μου παρέμβαση θα είναι ως συγγήτρια σε μια έκθεση για την τροφική αλυσίδα. Έφτασα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 20 χρόνια, εν μέσω της κρίσης των τρελών αγελάδων και αφού ήμουν υπεύθυνη για θέματα ε, τροφίμων και αγροτροφημικής βιομηχανίας στην Ισπανία. Στο μεταξύ δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ασφάλειας των Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, και ε, συμμετείχα ε, σε όλη την νομοπαρασκευαστική διαδικασία για την νομοθεσία της ασφάλειας τροφίμων. Έχουμε την πιο αυστηρή νομοθεσία για τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πρότυπο αναφορά σε θέματα επιστηστικής ασφάλειας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η βιομηχανία παραγωγή τροφίμων μα είναι εξαιρετική, καινοτόμα και ανταγωνιστική. Και η για την οποία είμαι σημείο αξιωματούχο επαφή, αρμόδια επαφή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Οργανισμό Αυτό Ασφάλεια Τροφίμων ασκεί με εξαιρετικό τρόπο το έργο τη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Βέβαια θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κανονισμό του 2002 για την ίδρυση του Οργανισμού Αυτού Ασφάλεια Τροφίμων. Όχι γιατί ο χρόνο έδειξε κάποια σημεία που επιδέχονται βελτιώσει, αλλά και γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτε όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για την διαδικασία προσδιορισμού του κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων και είναι υπέρ της διαφάνειας των επιστημονικών μελετών στις οποίες στηρίζεται η λήψη των αποφάσεων. Λυπάμαι όμως που πολύ σπευσμένα στη δική μας κοινοβουλευτική θητεία ε, προσπαθήσαμε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό και υπό τεράστια πίεση από τα ΜΜΕ. Αυτό ήταν πολύ αρνητικό. Και το να αποκαλούμε τον κανονισμό γενική νομοθεσία περί είναι λίγο στον φόδες και υπερβολικό, γιατί μόνο στο θέμα της διαφάνειας εγκύπτει. Α μην ξεχνούμε ότι το σύστημα ασφάλειας τροφίμων προβλέπει ευθύνη προσδιορισμού του κινδύνου για τις αρχές, τις αρμόδιες αρχές, αλλά όχι η διαχείριση του κινδύνου δεν εμπειρίπτει τι αρμόδιε αρχέ. Πιστεύω όμω ότι η συμφωνία μα είναι σημαντική. Πιστεύω ειλικρινά ότι υλοποίησαμε το στόχο μα, γιατί εξασφαλίσαμε μια διαδικασία λήψη αποφάσεων που στηρίζεται σε επιστημονικέ αποδείξει. Ε, Διασφυλάσσει υψηλό επίπεδο δημόσια υγεία και ασφάλεια στην Ευρώπη και πιστεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη στη λήψη αποφάσεων, γιατί καθιστούμε πιο διαφανή αυτή τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, οι πολίτες έχουν άμεση πρόσβαση στις επιστημονικές μελέτες που στηρίζουν τις αιτήσει ε, αδειοδότησης. Δηλαδή, οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται τη στιγμή της υποβολής, ε, ε, τη στιγμή της εξέτασης και της κρίσης της αίτηση ως παραδεκτής και έγκυρης. Και επίσης δημιουργείται βάση δεδομένων ώστε οι εταιρείε να υποβάλουν όλες τις επιστημονικές μελέτες όταν ζητούν άδεια και να μην υποβάλουν μόνο τις ευνοϊκές επιστημονικές μελέτες αλλά και τις αρνητικές. Και οι επιχειρήσεις που θα, δεν θα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις θα, θα για αυτές θα υποβάλλονται κυρώσεις. Πιστεύω ότι βρήκαμε ισορροπία μεταξύ της διαφάνειας και των συμφερόντων της βιομηχανίας, ώστε να συνεχίσουμε να τονώνουμε την καινοτομία στην ε, βιομηχανία παραγωγής τροφίμων της Ευρωπαϊκής, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάδοση των πληροφοριών θα γίνει υπό την επιφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων βιομηχανική ιδιοκτησία. Επίση, για να αποφύγουμε να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίε αυτέ για άδικου ε, εμπορικού σκοπού, προσθέσαμε και κάποιε ρήτρες ε, και ασφαλιστικέ δικλείδε ε, για την ε, δημοσιοποίηση της πληροφόρησης. Σε ό,τι αφορά την ΕΦΣΑ. Χαίρομαι για δύο λόγους. Από τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει δύο εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων και δεύτερον θα ε, παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις τεχνικές και επιστημονικές επιτροπές. Έτσι θα εμπλέκονται πιο στενά οι επιστήμονες από όλα τα κράτη-μέλη στις διαδικασίες χορήγησης άδεια. Σε ό,τι αφορά το κατάλογο με τα επιστευτικά στοιχεία, είναι σημαντικό η διαδικασία παραγωγής ή ε, παρασκευής να θεωρείται ως εμπιστευτικό στοιχείο. Επίσης, ε, οι καινοτόμε ιδέες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις εμπιστευτικές πληροφορίες, τα εμπιστευτικά στοιχεία. Άλλο θετικό στοιχείο είναι η αξιολόγηση του κινδύνου που θα στηρίζεται στις επιστημονικές αποδείξεις. Ταυτόχρονα θα βελτιώνεται η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Λυπούμε μόνο που δεν πιστοποιήθηκε η διαδικασία ε, ή δεν ε, ε, εξισώθηκε με την αντίστοιχη διαδικασία που ισχύει για, την, για τους οργανισμούς χημικών τροφίμων και φαρμάκων. Ευχαριστώ. Εξ ονόμα της Επιτροπής, το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος, κύριος Κατάινεν. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είναι υπερήφανη η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει το πιο αποτελεσματικό σύστημα για ασφάλεια τροφίμων και το πιο αποδοτικό στον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ταυτόχρονα ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τρόφιμα. Θέλουν να ξέρουν πού προέρχεται αυτό που τρώνε. Είναι κατανοητό ότι είναι ευαίσθητοι οι πολίτε μα για την αξιολόγηση του κινδύνου και τη διαχείριση του κινδύνου και τι σχετικέ αποφάσει στην αλυσίδα των τροφίμων. Άρα δεν θα σας εκπλήσει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν συμπληρωματικές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των τροφίμων τους. Τα πορίσματα της εφαρμογής των μέτρων και η πρωτοβουλία πολιτών η σχετική με τα διάφορα προβλήματα το έδειξαν αυτό. Πριν προχωρήσουμε να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το θετικό αποτέλεσμα τη διοργανική συζήτηση των πραγματεύσεων επί τη προτάσεω Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό περί διαφανεία και βιωσιμότητα του συστήματο ε, διαχείριση κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων είναι ένα σημαντικό βήμα. Και οι δύο συνομοθέτε έδειξαν ότι θέλουν να βρουν λύση για το θέμα αυτό έγινε ένας ε, επικοδομητικός, ανοιχτός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων. Καταφέραμε να φτάσουμε σε μια προσωρινή συμφωνία επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα δεκάμινο. Αυτή η προσωρινή συμφωνία για τους κανόνες περί διαφανείας Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι σημαντικός λίθος, ακρογωνίος λίθος για τις προσδοκίες των πολιτών που θέλουν περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων στην αλυσίδα τροφίμων. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποιες λεπτομέρειες, να αναφερθώ στα βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας και τους στόχους. Η προσωρινή συμφωνία αποτελεί αναθεώρηση του συστήματο ασφαλεία τροφίμων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω με σκοπό τη διαφάνεια, μεγαλύτερη διαφάνεια τη αξιολογήσεω του κινδύνου και της σχετικής διαδικασίας θα συμβάλλει στην νομιμοποίηση της ε, περί μεγαλύτερη νομιμοποίηση τη αρχή για την ασφάλεια των φήμων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγηση κινδύνων και η ΕΦΣΑ θα λογοδοτεί με καλύτερο τρόπο στους πολίτες. Έχοντας αυτό υπόψη, η προσωρινή συμφωνία προβλέπει την εθελοντική αποκάλυψη πορισμάτων των επιστημονικών μελετών ε, που τροφοδοτούν την επιστημονική ανάλυση. Αυτό γίνεται στην αρχική φάση της διαδικασίας αναλύσεως του κινδύνου από την στιγμή που έχει γίνει αποδεκτή μια αίτηση. Αυτή η αποκάλυψη στοιχείων συνδέεται στενά με δύο άλλες προτινόμενες ε, δράσεις, δημόσια διαβούλευση, υποβολή μελετών και κοινοποίηση των μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζουν το αίτημα αδειοδότησης και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο διαχειρίζεται η ΕΦΣΑ. Αυτά τα μέτρα θα εξασφαλίσουν ότι η ΕΦΣΑ μπορεί να έχει πρόσβαση στα επιστημονικά στοιχεία πριν να συντάξει τη δική της επιστημονική γνωμοδότηση. Η αυξημένη ε, διαφάνεια όσον αφορά το κοινό, έλεγχος του κοινού, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγηση του κινδύνου. Ταυτόχρονα αυτή η προσωρινή συμφωνία λαμβάνει υπόψη και άλλη ανάγκη. Να παραμείνει, να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ε, του τομέα ε, τροφίμων και ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσωρινή συμφωνία καθορίζει πάνω σε αυτό μέτρα διαφύλαξης για την ε, προστασία τεκμηριωμένων εμπιστευτικών πληροφοριών. Παρόμοια, η προσωρινή συμφωνία σέβεται υφιστάμενες διατάξεις για πνευματικά δικαιώματα, ε, προστασία των δεδομένων, των προσωπικών και δεδομένων που αφορούν τα προϊόντα που πρέπει να προστατευτούν. Όχι μόνο αυτό είναι κρίσιμο συστατικό που τονώνει την καινοτομία, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια αναγνώριση ευρωπαϊκών ε, προϊόντων και να αναγνωρίζεται η παγκόσμια ασφάλεια των ευρωπαϊκών προϊόντων. Για να βοηθήσουμε τους ετούντες και πιο σημαντικό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η προσωνή συμφωνία θεσπίζει τη δυνατότητα η ΕΦΣΑ να παρέχει συμβουλές πριν γίνει η αίτηση. Αυτή η συμβουλή θα διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση της διαδικασία υποβολής αιτήσεων και θα διευκολύνει τη ζωή για τις καινοτόμες εταιρείε. Για να εξασφαλίσουμε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ΕΦΣΑ, τα κράτη-μέλη θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ. Το Δικαιωτικό Συμβούλιο της ΕΦΣΑ συμπεριλαμβάνει και δύο μέλη που θα διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζουν τα αξιότιμα μέλη, αυτό είναι κάτι που αποκλίνει από την κοινή προσέγγιση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποκεντρωμένους οργανισμούς της 19ης Ιουλίου του 2012 θα διαβιβάσει δήλωση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εκφράσει τη λύπη τη για αυτή την παρέκκληση. Παρόμοια, και χωρίς να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ, τα κράτη-μέλη θα είναι πιο ενεργά στις διαδικασίες και θα εξασφαλίζουν την παρουσία εμπειρογνωμόνων στα επιστημονικά πάνελ της ΕΦΣΑ. Είναι σημαντικό λοιπόν να επισημένονται ε, οι κίνδυνοι και να κοινοποιούνται στου πολίτες. Η προσωρινή συμφωνία το αναγνωρίζει αυτό και σκοπεύει στο να βελτιώσει το σύστημα επικοινωνία των φάτους κινδύνους. Η συμφωνία δημιουργεί τα θεμέλια για πλήρη αποτελεσματική στρατηγική για την κοινοποίηση των κινδύνων. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το μήνυμα θα είναι σαφές, κατανοητό, ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ΕΦΣΑ ή από τα κράτη-μέλη. Προέδρε, αξιότιμα μέλη, σας επενώ για την ενεργό συμμετοχή σας, τη δραστηριοποίησή σας και την προσπάθεια που καταβάλλετε για να φτάσουμε στην προσθένη συμφωνία και προσβλέπω στα της, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κατάινεν. Εξ ονόματο της Επιτροπής Αλληλείας το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Σεράο Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ για το άρτιο έργο της, την εισηγήτρια και όλους όσους ενεπλάξαν στην εκπόνηση της έκθεσης. Λυπάμαι που δεν θα επικεντρωθώ τώρα στα άπειρα θετικά σημεία τη έκθεση, γιατί έχω μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μου. Θα ήθελα να σα προειδοποιήσω για το γεγονό ότι η παραγωγή τροφίμων από προϊόντα τη θάλασσα και των ωκεανών δυστυχώ δεν ε, τη χάνει τη μεταχείριση με την ε, γεωργική ή βιομηχανική παραγωγή. Και παρά τι ε, τροπολογίε που έγιναν, το, συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΣΑ, του Οργανισμού Ασφάλεια Τροφίμων, δυστυχώ δεν έχει κανένα εκπρόσωπο από την Αλία ή την εκθειοκαλλιέργεια ή την υδατοκαλλιέργεια. Ο τομέα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί περίπου 70% των προϊόντων που καταναλώνουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από προϊόντα αλληλεία ή υδατοκαλλιέργεια τα εισάγουμε από τρίτε χώρε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι και οι τρίτε αυτέ χώρε σέβονται τι ίδιε υψηλέ προδιαγραφέ ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων. Επίση, ζητούμε από του ωκεανού να συμβάλλουν σε μια πιο υγιεινή διατροφή. Σε ένα, στον πλανήτη μα, όπου η παχυσαρκία και οι παθήσει που οφείλονται σε αυτήν έχουν γίνει μια νέα μάστιγα με υψηλό κόστο και ευθύνονται για πολύ περισσότερου θανάτου από ό,τι θάνατοι λόγω λοιμού ή υποσυτισμού. Σα ευχαριστώ. Στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων και την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ντελαέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας ε, διαπιστώσαμε πως ε, τα θέματα που αφορούν τα φυτοφάρμακα και τη διαδικασία αδειοδότησης τους ε, είναι από τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τον Ευρωπαίο πολίτη. Θέλουν οι πολίτες να γνωρίζουν πώς λειτουργεί το ευρωπαϊκό σύστημα και είναι καθήκον μας ως αιρετοί και νομοθέτες να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών. Το συγκεκριμένο κείμενο ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στον προβληματισμό του πολίτη, καθιστά τις διαδικασίες πιο σαφείς και διαφανείς. Επίσης, ελπίζω ότι θα ε, αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους οργανισμούς μας και στις, ε, ε, στα νομοπαρασκευαστικά όργανα. Ο πολίτης θέλει περισσότερα στοιχεία δημόσια. Φυσικά θέλουμε διαφάνεια και στην επιστημονική έρευνα και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτού του ζητουμένου και της ανάγκης εξασφάλισης καινοτομίας οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις μας και η βιομηχανία μας αντιμετωπίζει το παγκόσμιο ανταγωνισμό. Θα πρέπει λοιπόν να τις επιτρέψουμε να διαφυλάξουν την πρωτοκαθεδρία του σε θέματα της καινοτομία. Χαιρετίζω το έργο της εισηγητρία τη κυρίας Πιλάρα Γιούσο και των σκιωδών εισηγητών. Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω στο τέλος αυτό της κοινοβουλευτικής θητείας ε, την επιθυμία μου οι αποφάσεις που λαμβάνομαι να δράζονται πάντα σε στέρεες επιστημονικές βάσεις και αποδείξεις. Μόνο έτσι θα έχουμε τα κριτήρια και θέσεις για να μην τροφοδοτούμε τον ε, φόβο για τα τρόφιμα που μερικές φορές κάποιοι εκμεταλλεύονται για κομματικούς ή ψηφοθερικούς σκοπούς. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών μας και ιδίω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Είναι σημαντική η σωστή λειτουργία τέτοιων οργανισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντάλη, ανάμεσα των Σελιστών έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι θυμόμαστε το σκάνδαλο με τις πιέσεις της χημικής βιομηχανίας για να εγκριθεί η γλυφοσάτη στα ζυζανιοκτώνα και βεβαίως ε, η απάντησή μας ήταν η ενδεδειγμένη και νομίζω ότι αυτό δείχνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η φωνή των πολιτών.